Συνεχίζουμε με την ημερησία διάταξη. Περνάμε στις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το πολιετές πρόγραμμα 2010-2014 σε σχέση με το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Έχει τον λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου η κυρία Άσκ παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε